Okay, ladies and gentlemen, let's start. Äh, Σας äh, καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί έχουμε τρία ε, θέματα στη μεσία διάταξη, τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε μαζί. Ε, το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. έχουμε ε, την, ε, διάφορες δραστηριότητες στο πρόγραμμα πλαίσιο ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Ο συνάδελφος Πρεζίνα έχει αναλάβει το θέμα και θα τον παρακαλούσα να πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει το θέμα. Κατόπιν θα περάσουμε στην κοινή συζήτηση. I'm sorry, Mr. Uh, Mr. Já Θα ήθελα εκ μέρου ε, ολόκληρη τη επιτροπή μα, θα ήθελα να ευχηθώ στον πρόεδρό μας χρόνια πολλά. Γιατί ο καταπληκτικός μας πρόεδρος σήμερα έχει γενέθλια. Θα ήθελα λοιπόν να του ευχηθώ σιδερένια υγεία, μακροημέρευση και είναι σημαντικό όταν κανείς γίνεται 18 χρονών και είναι τόσο σοφός να το γιορτάζει. Σας ε, ευχαριστώ θερμά. Ήλπιζα ότι δεν θα, ότι δεν θα φαινόταν ότι έχω ε, ε γεράσει. Ε, και ότι δεν το πρόσεχε κανείς. Έπασε τόσο, ο κύριος Μπεζίνα έχει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά από ό,τι είχα προγραμματίσει. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση στις 7 Μαρτίου του 2011 η Κομισιόν υπέβαλε ε, το πακέτο με νομοθετικές προτάσεις ε, για την εκπαίδευση στον ε, τομέα της ατομικής ενέργειας για τα χρόνια 2012 με 2013. Είναι συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία προβλέπουν ε, έμεσες και άμεσες δράσεις. Ε, προβλέπεται και η συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο. Πολύ σύντομα μπορούμε να πούμε ότι οι προτάσεις του προγράμματος πλαισίου για τα έτη 2013 2012 ε, και 2013 υπάρχουν επειδή ο κύκλος πάντα διαρκεί 5 χρόνια, τα, η διάρκεια των προγραμμάτων όμως είναι 7 χρόνια και γι' αυτό ε, έχουμε πάντα αυτά τα δύο χρόνια όπου θα πρέπει να κάνουμε κάποιο γεφύρωμα. Και ε, η έρευνα που χρηματοδοτείται από ε, το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα και για την χρήση της ατομικής ενέργειας στη βιομηχανία και στη γιατρική. Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα συνδέονται και με την Ευρωπαϊκή ε, πρωτοβουλία για την ε, βιώσιμη ε, πυρηνική ενέργεια. Πρόκειται για μία από τις έξι βιομηχανικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τεχνολογίες ενέργειας. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, σχετικά με ε, την χρήση της ε, ατομικής ενέργειας. Το ερώτημα της χρήσης ή μη αυτής της ενέργειας είναι κάτι που αναπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα ε, στην ατομική ενέργεια. Μετά την ε, Φουκουσίμα η Ευρώπη ε, πρέπει να προσέξει περισσότερο την ατομική ενέργεια, πρέπει να κοιτάξει την ασφάλεια, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και να εξετάσει και το ενδεχόμενο της σύνδεξης. Είναι θέματα αυτά τα οποία βίπτουν ε, στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ε, πρέπει όμως ε, να φροντίσουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Με την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας μπορούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία, διότι θα ήθελα να τονίσω Ε, ότι δεν συμμερίζεται όλη η Ευρώπη την απόφαση ε, να εγκαταλείψει την ε, πυρηνική ενέργεια. Οι έρευνες λοιπόν πρέπει να συνεχίσουν. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ επίκαιρη. Κάποια ερευνητικά κέντρα όπως για παράδειγμα αυτό στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εξασφαλίσει την ε, χρηματοδότησή τους μόνο μέχρι το τέλος ε, του χρόνου. Ε, για να υπάρξει λοιπόν συνέχεια στις έρευνες θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο χρόνια. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση και προσλέπω στην συνεχιζόμενη συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι πολύ σύντομε οι προθεσμίες ε, στη συνέχεια του χρονοδιαγράμματος και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 6 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ε, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή. Δεν ζητάει κανεί το λόγο. Η κυρία Χέρτσοκ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, γιατί πέρασε όλες του τις θερινές διακοπές με τις εκθέσεις αυτές. Γιατί πραγματικά είχαμε πολύ στενό χρονοδιάγραμμα και αφιέρωσε όλο τον ελεύθερο χρόνο σε αυτό. Τον συγχαίρω λοιπόν και τον ευχαριστώ. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να δουλεύει κανείς ε, μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά στην περίπτωση αυτή είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα γιατί φαίνεται ότι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο αλλά ίσως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν και θέλουν μάλλον να γεφυρώσουν ε, ε, ένα χρονικό και δημοσιονομικό χάσμα παρά να λάβουν μια μεγάλη επίβολη πολιτική απόφαση για τα πυρηνικά. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και η γνωμοδότησή μας αυτή έχει μάλλον δημοσιονομικό χαρακτήρα, αφορά τον προϋπολογισμό παρά οτιδήποτε άλλο. Και οι περισσότερες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούν να συνδυάσουν τον ε, προϋπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με το ερευνητικό πρόγραμμα της Euratom. Αυτό, αυτός είναι ο σκοπός μας, να μην χάσουμε ενέργεια στις συζητήσεις για το θέμα αυτό, αλλά να βελτιώσουμε την κατάσταση πιστεύω ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες, τουλάχιστον οι δικοί μας, έχουν αντιληφθεί ότι αν γίνουν ρηξικέλεθες αλλαγές στο θέμα των πυρηνικών, η έρευνα θα πρέπει να ενισχυθεί σε ορισμένους τομείς. που είναι σημαντική. Χρειαζόμαστε λοιπόν και κονδύλια και για να εξασφαλίσουμε τα μέσα αυτά, τα οικονομικά για την έρευνα και τους νέους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας θα πρέπει να ε, δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα, στην εξασφάλιση των κονδυλίων. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες με στόχο να αναφέρουμε αυτούς τους ε, δυνάμει σημαντικούς τομείς της ε, πυρηνικής έρευνας, όπως είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας, και στόχος μας είναι η Επιτροπή μας σύσσωμη να στηρίξει την έκθεση και να εξασφαλίσει τους απαραίτητους χρηματοπιστωτικούς πόρους. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά συνενετική γνώμη. Αυτό προσπάθησε ο κύριος Μπρεζίνα με τις εκθέσεις του και πραγματικά το έργο του είναι αξιέπαινο. Και να δούμε τι θα γίνει και στο Συμβούλιο να εξετάσουμε τις προτάσεις του Συμβουλίου και να τις ε, ενσωματώσουμε ίσως και στη δική μας έκθεση για να έχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε και μάλλον υπάρχει συνένεση. Ευχαριστώ κύριος Μετζάρος. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και ο συνάδελφος μίλησε τσεχικά, να μιλήσω κι εγώ σλοβακικά για να με καταλάβει καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον κύριο Μπρεζίνα, για το πολύ αξιόλογο έργο του. Το θέμα της πυρηνικής έρευνας θα πρέπει να βρεθεί πραγματικά στο επίκεντρο του προβληματισμού μας μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα και μετά τα πολλά σημεία και τα προβλήματα που ανέκυψαν καθώς και τις ανησυχίες που προέκυψαν μετά τη Φουκουσίμα. Είδαμε και τις αντιδράσεις ε, πολλών χωρών και περιμένουμε τη μελλοντική του στάση σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια. Συμφωνώ με τον κύριο Ψέζινα ότι χρειάζεται ε, μετά τη Φουκουσίμα να ενισχύσουμε, να επιτείνουμε την ε, έρευνα στα πυρηνικά και όχι να την μειώσουμε. Θα πρέπει να διδαχθούμε από το μάθημα της Φουκουσίμα και να το χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία για να επισημάνουμε την ανάγκη περισσότερης έρευνας ε, στον πυρηνικό τομέα. Και στα πλαίσια του 8ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε διάφορους τομείς πυρηνικής έρευνας. Και όπως είπε και η κυρία Χέρτσοκ, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα απαραίτητα κονδύλια, τα οικονομικά μέσα για να χρηματοδοτήσουμε τα ερευνητικά μας σχέδια και προγράμματα. Ε, ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι η ασφαλής ε, αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων ή η ασφαλής μεταφορά πυρηνικού υλικού. Όλα αυτά τα θέματα θα μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο της μελλοντική έρευνας για τα πυρηνικά. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν την εμβάθυνση αυτής της έρευνας και επίσης ένα μακροπρόθεσμο ερευνητικό πρόγραμμα δεν θα πρέπει να παραμελεί το θέμα της σύνδεξης. Το πρόγραμμα ITER δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο των προτεραιοτήτων μας. Πάντω, δεν νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μα στα πυρηνικά. Το αντίθετο θα πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σίζελ. Ευχαριστώ. Οι επενδύσει στην ενέργεια, στην πυρηνική ενέργεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι τελευταίε τρει δεκαετίε ήταν πολύ οι επενδύσεις ήταν πολύ χαμηλές. Ε, το ίδιο και οι επενδύσεις στην έρευνα. Δεν έγιναν επενδύσεις ούτε στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησαμε ότι ε, δεν είναι δεδομένη η ασφάλεια του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού και τότε αρχίσαμε να εξετάσουμε πιο σοβαρά την πιθανότητα επένδυσης και στην πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε από τη μια να είμαστε κατά μιας μορφής ενέργειας και από την άλλη να θεωρούμε ότι είναι αυτή η πηγή ενέργειας μια ασφαλής ενεργειακή πηγή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει κάπως το κλίμα που επικρατεί για την πυρηνική ενέργεια και νομίζω ότι Εκεί επικεντρώνονται και οι δικές μας προσπάθειες. Πιστεύω ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι απαραίτητο στοιχείο της όλης προσπάθειας και συμφωνώ απόλυτα με τις ε, εκθέσεις του κυρίου Ψέζινα και θα ήθελα να το συγχαρώ. Πρέπει να δώσουμε μία σωστή απάντηση στο πρόβλημα της Φουκουσίμα. Θέλουμε έρευνα που δεν θα εξασφαλίσει μόνο το ισχύον επίπεδο προστασίας και ασφάλειας, αλλά θα το ενισχύσει. Επίσης, στην Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε και πιο οραματιστές, ώστε να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά τις πηγές ενέργειας για την παραγωγή ενέργειας. Και δεν θα πρέπει να χάνουμε και την αισιοδοξία μας για τη σύνδεξη. Ας μην ξεχνάμε ότι η πυρηνική ενέργεια δημιουργεί και απόβλητα και θα πρέπει να φροντίσουμε για την ασφαλή επεξεργασία τους ή αποθήκευσή τους. Η ανακύκλωση των πυρηνικών αποβλήτων είναι ένας τομέας που θα μπορούσε να βρεθεί ε, στο επίκεντρο της έρευνας για τα πυρηνικά. Και το θέμα του των ανθρώπινων πόρων είναι σημαντικό και έχουμε σχετική τροπολογία του εισηγητού. Εξετάζοντας τους κινδύνου τη πυρηνική ενέργεια, διαπιστώνουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πιο σημαντικός ε, και βαρύνει πιο πολύ στον κίνδυνο από ότι ο τεχνολογικός παράγοντας. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε και στην ε, διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση και του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού. Εγώ πιστεύω ότι η πυρηνική ενέργεια θα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό του ενεργειακού μείγματο με βάση τα έγγραφα στρατηγικής μας, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην πυρηνική ασφάλεια. Και αυτό το θέμα χρήζει ενισχυμένης χρηματοδότησης, γιατί η πυρηνική ασφάλεια, ιδιαίτερα μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, χρήζει ε, βελτίωσης και ενίσχυσης. Συμφωνώ με την συνάδελφο Χέρτσοκ που το επισήμανε. Σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο, πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η ευθυγράμμιση του χρονοδιαγράμματος της έρευνα της έκθεσης αυτής με το χρονοδιάγραμμα εκθέσεων για άλλα σημεία στρατηγικής. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια στρατηγική συνέχεια αυτού του προγράμματος. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους οι οποίοι υποστηρίζουν την πρόταση και θα συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή. Έχει έλθει πλέον η στιγμή κατά την οποία η συζήτηση των πυρηνικών θεμάτων έχει καταστεί κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο μετά από το συμβάν της Φουκουσίμα. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Μπρεζίνα κατάφερε να παρουσιάσει μια πολύ καλή έκθεση. Συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα είπαν σωστά πράγματα και δεν θα τα επαναλάβω. Επαναλαμβάνω πάντως την άποψη ότι η έρευνα θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται. Η καταστροφή της Φουκουσίμα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σημάνει το τέλος της πυρηνικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας κάθε τραγωδία και κάθε καταστροφή οδήγησε στους ανθρώπους να βγάλουν στα κατάλληλα συμπεράσματα και να αναζητήσουν το τι πήγε άσχημα. Πάρα πολλές καταστροφές και πάρα πολλές τυχίες ε, μας οδήγησαν στο να μάθουμε από τα λάθη μας και πολλές φορές οι καταστροφές στην ουσία έδωσαν όθηση στην τεχνολογική ανάπτυξη. Όσο πιο περίπλοκη είναι η τεχνολογία, τόσο πιο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κανείς τα επικίνδυνα θέματα όπως την πυρηνική έρευνα. Γι' αυτό χρειάζεται η πυρηνική έρευνα έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η ασφάλεια στον πυρηνικό τομέα είναι πολύ περισσότερη από οποιοδήποτε άλλο τομέα. <laughs> Και η πυρηνική ακριβώς ε, ενέργεια μπορεί να μας μάθει πάρα πολλά χρήσιμα. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει το ίδιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έρευνα και τότε μόνο θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας στον συγκεκριμένο τομέα. Να πω λίγα πράγματα τώρα να μου επιτρέψετε για το ΙΤΕΡ. Όπως μας είπε ο εισήγητής, η σύνδεξη είναι η μία από τις διαστάσεις της πυρηνικής έρευνας. Νομίζω ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να προχωρήσει η έρευνα σε πραγματικό επίπεδο. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι καλύτερη διαχείριση. Πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση οδεύουμε και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να γνωρίζουν σωστά και το χρονοδιάγραμμα για την έρευνα. Πολλοί από εμά έχουν εμπειρίες είτε πανεπιστημιακού είτε ερευνητικού τύπου και μερικές φορές παρουσιάζεται ο κίνδυνος η έρευνα να είναι αυτός Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ε, χρονοδιαγράμματα πάρα πολύ μεγάλα όπως στην περίπτωση του Ίτερ, που μας ανησυχούν. Δεν λέω ότι είναι αυτός η έρευνα για το Ίτερ, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα παραμείνει προς τη σωστή κατεύθυνση, να πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η συνάδελφος που πήρε το λόγο πριν από μένα αναφέρθηκε στην σημασία την οποία έχει η συνέχιση εκπαίδευσης πυρηνικών εμπειρογνωμόνων. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πάντα θα είναι διαθέσιμη η εμπειρογνωμοσύνη τους γιατί η πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει σημαντική στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία αν είναι της μόδας ή όχι η ενέργεια αυτή. Αυτό το οποίο χρειάζεται όμως είναι σωστά εκπαιδευμένοι εμπειρογνώμονες. Εμείς πρέπει να εξηγήσουμε την ανάγκη αυτή και να πάρουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να μην χάσουμε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη. Υποστηρίζω λοιπόν την έκθεση Μπρεζίνα και συγχαίρω τον κύριο Μπρεζίνα για μια εξαιρετικά ισορροπημένη ε, δουλειά την οποία έχει επιτελέσει. Μέσω της συζήτησης μπορούμε να βελτιώσουμε ένα ήδη εξαιρετικό έγγραφο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χίπνερ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και, τους, ε, και τον συνάδελφο για την ε, πολύ οξυδερκή του έκθεση θα εξετάσουμε την έκθεση και είδαμε και τις τροπολογίες. Φαίνεται ότι όλες οι πλευρές ε, ασχολήθηκαν με τη δέουσα προσοχή και έδειξαν τον ΔΕΟ ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Πολύ συχνά η κοινωνία φαίνεται δεν γνωρίζει τι σημαίνει για μας η πυρηνική ενέργεια και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να την θυσιάσουμε. Χαίρομαι που δεν ακούσαμε εδώ καμία φωνή που να λέει να κλείσουμε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς και να απελευθερώσουμε την Ευρώπη από την πυρηνική ενέργεια. Γιατί στην αρχή αμέσως μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα ακούστηκαν και κάποιες τέτοιες φωνές. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πιο σημαντικό πράγμα για μας, δηλαδή ε, ζητούμε ενίσχυση της πυρηνικής έρευνας. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, εμβάθυνση και διεύρυνση της έρευνας για τα πυρηνικά. Αυτό είναι το ζητούμενο και ο εισηγητής μίλησε και για την ασφάλεια. Ε, στην Φουκουσίμα το πρόβλημα δεν ήταν η τεχνολογία, αλλά τα συστήματα αυτοματισμού και σε αυτό θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Με τις έρευνες, με περισσότερες μελέτες, με επικουρικά συστήματα ασφάλειας, να ε, συμπληρώσουμε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις ε, έρευνες για τα πυρηνικά και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να τις χρηματοδοτήσουμε. Δεν αρκεί μόνο να μιλάμε για το θέμα αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και χρηματοοικονομική υποστήριξη. Αλλιώς με τα ωραία λόγια δεν πρόκειται να σημειώσουμε καμία πρόοδο στην έρευνα και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Πολύ σωστά ο εισηγητής αναφέρθηκε στο θέμα των αποβλήτων, όχι μόνο ε, στο θέμα της μεταφοράς των αποβλήτων και της ε, αποθήκευσης, αλλά μίλησε για έρευνες και στα θέματα τεχνολογίας απομπλουτισμού των αποβλήτων, ώστε να γίνουν πιο ουδέτερα για το περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα είδος εξουδετερώσης ε, των αποβλήτων από, τις πυρηνικ... από τους πυρηνικούς σταθμούς ή ουδετεροποίησης. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η πληροφορία προς τον κόσμο, προς το κοινό. Εκεί είναι που χάνουμε, γιατί ο κόσμο είναι πεπισμένο ότι η πυρηνική ενέργεια, η ατομική ενέργεια είναι η χειρότερη πηγή ενέργεια. Αυτό δεν ισχύει. Είναι λαθασμένη αντίληψη. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ενημέρωση προ του πολίτε γιατί μέσω στη ενημέρωση και την υποστήριξη της έρευνας μπορούμε με αξιόπιστο τρόπο να παρουσιάσουμε και αντικειμενικά στους πολίτες ε, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ατομική ενέργεια. Και στο θέμα της και στο θέμα της ε, ενημέρωσης των πολιτών θα πρέπει να προβλέψουμε απαραίτητα κονδύλια. Και απευθύνω μία έκκληση προς τους συναδέλφους ε, των διαφόρων χωρών. Δεν πρόκειται να αποφύγουμε τη δημόσια συζήτηση, την κοινωνική συζήτηση για τα πυρηνικά. Γι' αυτό όσο πιο γρήγορα αναμειχθούμε σε αυτή τη συζήτηση και όσο πιο γρήγορα ε, προσφέρουμε στους πολίτες αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο πιο εύκολη θα είναι η συζήτηση. Γιατί αυτό περιμένει από μας ο κόσμος, αυτό περιμένει από μας η κοινωνία, ώστε να διασκεδαστούν οι φόβοι. Θα πρέπει να δώσουμε έγκαιρα τις πληροφορίες για να διασκεδαστούν οι αφιβολίες ότι η ατομική ενέργεια είναι πραγματικά μια ασφαλής μορφή ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σαν πράσινη γύρω από την έκθεση αυτή γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις προτεραιότητες οι οποίες ακούστηκαν. Υπάρχουν 453 πυρηνικοί αντιδραστήρες στον κόσμο πριν να κλείσουν οι γερμανικοί αντιδραστήρες και εδώ και 25 χρόνια υπέστη με το Τσέρνομπιλ, τη Φουκουσίμα πριν λίγους μήνες και δεν μπορούμε να πούμε ότι η ασφάλεια είναι απόλυτη. Να πούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για την ασφάλεια, φυσικά ας δώσουμε εγγυήσει. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τις υπεργολαβίες γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν οκτώ κλίμακες υπο, υπο, υποεργολαβίας που ε, είναι κάτι που φύγει την ασφάλεια στη διαχείριση των αντιδραστήρων είτε στη Γαλλία είτε αλλού. Και ας ενισχύσουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις μετά από τα stress test έγιναν ορισμένες αξιολογήσεις και χρειάζονται περίπου ένα δις ευρώ ανά πυρηνικό ε, αντιδραστήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ε, κάλυπτρα τσιμεντένια με ενίσχυση γύρω από τις ε, γεννήτριες κτλ. Σήμερα στο κανάλι Ανσενέ λέγεται ότι όταν κατασκευάζουμε μια τέτοια εγκατάσταση διαπιστώνουμε ότι το ενισχυμένο τσιμέντο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι υπονομιβμένο και είναι πρόβλημα λοιπόν και ο βομβαρδισμός με το ουράνιο των προϊόντων αυτών δημιουργούμε προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν σε σχέση ε, με το περιβάλλον. Μιλάτε τώρα για την τέταρτη γενναία η τέταρτη γενεά λειτουργεί και αυτή με την ίδια μέθοδο, πως το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Και μετά λέτε, α ωραία τώρα έχουμε τη σύνδεξη. Εν πάση περιπτώσει είχαμε πάει στο Κανταράς κάποιοι από εμά. Και η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τεράστια επιστημονικά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Και δεν συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πούμε ότι θα, πούμε, ότι θα επενδύσουμε ε, το 2006 5 δις, τώρα είμαστε στο 11 και έχουμε επενδύσει 15 δις και πάντα έχουμε ερωτηματικά γιατί το κάλυμα αυτή της συγκεκριμένης ε, ε, εγκατάστασης είναι αντικείμενο πειραματισμών στο JET στην Μεγάλη Βρετανία και τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει γνωστά και με το ITER λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα JET στην Μεγάλη Βρετανία και μετά θα δούμε τι να κάνουμε. Ας παγώσουμε τα πράγματα. Ενώ τώρα θέλετε να ξοδέψετε ευρωπαϊκές πιστώσεις για αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν 100 χρόνια μετά. Σας κάνω μια πρόταση κύριε Σιγητή. Αυτό που είπε η προηγούμενη συνάδελφος, βελτιώστε την ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος της Φουκουσίμα, Υπάρχουν χιλιάδες ε, σένσορες στον υπόλοιπο κόσμο που ανοιχνεύουν τα σύννεφα που δημιουργούνται από τη Φικουσίμα. Και αυτό το διεθνές δίκτυο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ε, απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών, λέγεται CBCT και είχε όλα τα αποτελέσματα αναώρα για την κατάσταση σε ε, εξένιο, σε κέσιο, αναώρα και τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Η πρόταση η οποία κάνω λοιπόν είναι να βελτιώσουμε την ενημέρωση γιατί η υποχρέωση του να υποστούμε τις συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης μας δίνει το δικαίωμα να γνωρίζουμε. Και ακριβώς αυτή η συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων Ας ζητήσουμε τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από την απόφαση αυτή να είναι δημόσια. Γιατί θα πρέπει να περιμένει κανείς και άλλα ατυχήματα. 453 πυρηνικοί αντιδραστήρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ασφάλειας, γιατί το ατύχημα συμβαίνει επειδή δεν το προβλέψαμε. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι λοιπόν εμείς και ο πληθυσμός, γιατί μέχρι τώρα μόνο τα κράτη και μόνο αυτοί που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση αυτή. Πρέπει η πληροφόρηση αυτή να είναι δημόσια, είναι μια ξεκάθαρη, ε, ε, είναι ένα ξεκάθαρο αίτημα αυτό το οποίο κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η διεθνής ε, συνεργασία πιστεύω θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον και γι' αυτό η ενισχυμένη ε, συνεργασία με την ε, Διεθνή Αρχή Ατομικής Ενέργειας επίσης είναι σημαντική και θα είναι καλό να τεθούν ε, υποχρεωτικά πρότυπα ώστε να μπορούν να γίνονται έλεγχοι από ε, ε, επίσημους επιθεωρητές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει και την απαραίτητη κατάρτιση. Με την συζήτηση περί Ιαπωνίας ε, συζητιέται περισσότερο η διάθεση των αποβλήτων. Θα πρέπει να γίνουν ε, μεγάλες προσπάθειες ε, διότι όλο αυτό θα σημάνει και σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Όσον αφορά το ίτερ, θα ήθελα να πω ότι φυσικά θα πρέπει να τηθούν οι διεθνείς ε, συμφωνίες. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι ε, μέχρι το 2020, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διεθνείς ε, συμφωνίες. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον Μπεζίνα. Έχει κάνει μια τεράστια συνθετική δουλειά σε μια πάρα πολύ δύσκολη, ε, σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Ακούσαμε τις απόψεις των πρασίνων, πράγματι κάνουμε έναν κατάλογο των ατυχημάτων και προωθούμε τον φόβο. Αυτό θα έλεγα μου θυμίζει ε, την αντίδραση ε, των κατοίκων της Στύλου όταν δημιουργήθηκε το τρένο γιατί φοβόντουσαν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό τους ότι ε, θα φυγούν από αυτό και τώρα η πόλη της Μπρίβ Λαγκαγιάρντ πήρε τον τελικό σταθμό και τη γραμμή του τρένου και έχει αναπτυχθεί τρεις φορές περισσότερα από την πόλη της Τούλ. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβόμαστε την επιστήμη σε τέτοια σημαντικά θέματα όπως η ενέργεια. Ε, συγχαίρω την Επιτροπή για την πρότασή της, γιατί πράγματι αναφέρεται σε επιστημονικά θέματα. Για το ίτερ μιλήσαμε πάρα πολύ για τα δημοσιονομικά και επιτέλους ένα συνάδελφος είπε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και πρέπει να στηρίξουμε τη μέθοδο της σύνδεξης. Δεν, μια δεύτερη παρατήρηση, είχα κάνει παλιά την πρόταση για το κοινό κέντρο έρευνας να του ζητήσουμε ένα πρόγραμμα για την διάλυση των παλαιών μονάδων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Έχουμε εξαιρετικούς μηχανολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει να εφόσον έχουμε τους καλύτερους ειδικού στον κόσμο για τη διάλυση των εγκαταστάσεων να το εκμεταλλευτούμε. Πράγματι η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων για 100 ας πούμε χρόνια το πρόβλημα της διάλυσης των εγκαταστάσεων αυτών τίθεται. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Μία παρατήρηση για τη γραμματεία τώρα. Στο έγγραφο λέγεται ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει. Εμείς δεν εγκρίνουμε, γνωμοδότηση δίνουμε. Δεν έχουμε πολιτική αρμοδιότητα για την Ευρατών, τη συνθήκη Ευρατών. Ευνοϊκή, αν θέλετε, σύσταση, γνώμη, ό,τι θέλετε. Όχι όμως αποφασίζει. Θα σημειώνουμε αυτά, θα, θα το ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό. Συνάδελφος Ρέμεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμηση και το θαυμασμό μου για το έργο του εισηγητού μας Γιάννη Ψεζίνα για τις ατέρμονες συζητήσεις περί ενέργειας, ενεργειακού μείγματος και τη θέση της πυρηνικής ενέργειας σε αυτό το μείγμα. Μετά τη Φουκουσίμα η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ την πυρηνική έρευνα και θα πρέπει να διατηρήσουμε το ισχύων επίπεδο και ανθρώπινων πόρων και δεξιοτήτων εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας. Δεν είναι ότι τώρα επειδή κάποια κράτη-μέλη γύρισαν την πλάτη στην πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να μειώσουμε τις προσπάθειές μας στην πυρηνική έρευνα. Συμφωνώ με τον εισηγητή για τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και την ανάγκη της επικέντρωσης της έρευνας στα θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και την έρευνα για την πυρηνική σύνδεξη, γιατί άλλη επιλογή δεν έχουμε, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να βρούμε πηγές ενέργειας και θα ήταν πολύ κοντόφθαλμο αυτή τη στιγμή να κλείσουμε ή να τερματίσουμε το πρόγραμμα ITER μόνο και μόνο επειδή ο ορίζοντάς του είναι μακροπρόθεσμος και μερικοί από εμά δεν θα προλάβουν ε, να δουν τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Θα ήθελα ταυτόχρονα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ρόλο που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα πυρηνικής έρευνας. Και συμφωνώ ότι η γεωργία, η βιομηχανία και τα νοσοκομεία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή πυρηνικών αποβλήτων και όχι μόνο η πυρηνική σταθμή και τα πυρηνικά εργοστάσια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στην Κομισιόν στον κύριο Στρόμαϊερ ε, και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Πρεζίνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Ε, θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την ε, προσοχή του Κοινοβουλίου στο γεγονός ότι κατά την προετοιμασία της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου και μιλώ υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου, είναι παρόν εδώ το Συμβούλιο, ε, έγινε σαφές ότι κάποιες αντιπροσωπείες ήταν πολύ επιφυλακτικές, ε, για να το πω ήπια, να δεχτούν αναφορές ε, στην ανάπτυξη μελλοντικών συστημάτων. Ίσως λοιπόν θα θέλατε να σκεφτείτε μήπως όλες τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με αυτόν τον νέο τύπο εγκαταστάσεων Μήπως η συμπερίληψη των ε, τροπολογιών αυτών ε, θα ήταν αντιπαραγωγική ε, κατά την συζήτηση του, της έκθεσης με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και όλες τις τροπολογίες που συνδέουν το θέμα αυτό με τα προβλήματα στο ίτερ που θα πρέπει να λυθούν. Και όσον αφορά την ε, παρέμβαση της κυρίας Αγκάζη, θα ήθελα να πω ότι την ε, προηγούμενη εβδομάδα το ΤΣΕΤ ε, έχει παράγει πλάσμα τέτοιου τύπου, το οποίο φαίνεται να είναι και καλή ποιότητα. Σε, σε απάντηση λοιπόν της παρέμβασης αυτής θα ήθελα να πω ότι από το ΤΣΕΤ έχουμε ε, κάποια πρώτα αποτελέσματα. Επίσης θα ήθελα τέλος ε, να ενθαρρύνω το Κοινοβούλιο να ε, ε λάβει προορατική στάση όσον αφορά και τον φάκελο 7 συν 2 συμπεριλαμβανομένου του φακέλου ΙΤΕΡ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο, εισή, ο εισηγητής, ο κύριος Μπρεζίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις σας και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω την ανάγκη χρηματοδότησης που επισήμανε η κυρία Χέρτσοκ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της πυρηνικής έρευνας και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα απαραίτητα κονδύλια. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι και η ανθρώπινη πόρη είναι σημαντική. Ο κυρία Σιζέλη, ο κύριος Μεσάρος αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Και είναι γεγονός ότι στην περίπτωση Twitter πολύ συχνά προσκρούμε στην, ε, σε μια δυναμία διαχείρισης τέτοιων μεγαλεπίβολων σχεδίων. Αυτό επισήμανε ο κύριος και ότι είναι μερικές φορές αποτρεπτικός ο μακροπρόθεσμος χρονικός παράγοντας, ορίζοντας. Η κυρία Χιούμπνερ μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης ε, της επικοινωνίας μας με τους πολίτες προκειμένου να εξηγήσουμε καλύτερα τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας. Στην κυρία Ριβάζη θα ήθελα να πω ότι και εγώ ήμουν υπέρ της α, μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και ιδιαίτερα σε περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων και σε ό,τι αφορά την έκκληση στην ατμόσφαιρα στοιχείων όπως ο Κέσιο και άλλα που είχαμε με τη Φουκουσίμα θα πρέπει να έχουμε πλήρη διαφάνεια ε, του ελέγχου και της ε, παρακολούθησης της κατάστασης. Είμαι κατά οποιοδήποτε οποιοδήποτε περιορισμού όμως σε θέματα πυρηνικής έρευνας. Και θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι γνωρίζω πως μερικές αντιπροσωπείες δεν θέλουν να περάσουν στην επόμενη γενιά, στην τέταρτη γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων, αλλά εγώ επιμένω ότι η έρευνα δεν θα πρέπει να περιοριστεί και να μην καλύψει και θέματα αντιδραστήρων τέταρτης γενιάς. Κύριε Ρούμπιχ, σε μία τροπολογία μου μιλώ για την βελτίωση της συνεργασίας με την Διεθνή Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας. Πολύ σωστά ο κύριος Οντί υπέβαλε κάποια σχόλια και μια και η διορία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ σύντομη, βραχία λίγη στις 6 Σεπτεμβρίου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δημονώ για την συνέχιση της συνεργασίας με τους σκιώδεις σύγητες και ελπίζω ότι θα αξιοποιήσουμε τις διάφορες προθεσμίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση τη πυρηνική έρευνα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ähm, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρεζίνα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω Τις ε, προθεσμίες τις έχουμε ήδη αναφέρει, είναι πολύ σύντομες, έχουν όμως συμφωνηθεί. Αυτό είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί γρήγορα το ζήτημα. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους ε, να συνεργαστούν ώστε να τηρήσουμε τις ε, προθεσμίες. Ο κύριος Πρεζίνα έχει κάνει πολλή δουλειά στις διακοπές, έτσι έχει ήδη προωθήσει κάπως το θέμα, ε, ώστε να ολοκληρωθεί το θέμα εγκαίρως. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο το κεφάλαιο αυτό. Ε, είναι φορτισμένο θέμα πολιτικά. Ε, είμαι βέβαιος όμως ότι θα καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά και κλείνω το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Όχι, δεν περνάμε ακόμα, διότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 10. Μικρό διάλειμμα, σύντομο διάλειμμα. Πάρτε μια ανάσα και στις 10 ακριβώς θα συνεχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Yeah. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ την προσοχή σας. Ο κύριος Κάνον θα ήθελε να μας κάνει μια ανακοίνωση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. λυπούμε πω το λόγο για ένα τόσο ίσονο σημασία πρόβλημα, αλλά έχω ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο της φωνής και την ένταξη. Η διερμηνία είναι καταπληκτική, δεν παραπονιέμαι γι' αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά είναι πολύ χαμηλό, χαμηλή, χαμηλός ο ήχος. Χρειάζεται να βάλω στο, τον ήχο στο πιο δυνατό. Και μετά ακούω πολύ δυνατά αυτούς που μιλάνε. Ε, πραγματικά θα χάσουμε την, ε, την ακοή μας σε λίγο. Δεν θα ήθελα να χρειαστεί να μηνύσω μετά από λίγα χρόνια το κοινοβούλιο επειδή θα έχω κουφαθεί. Γι' αυτό παρακαλώ βοηθήστε με, ας κάνουμε κάτι. Ε, όχι, πραγματικά δεν ε, μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Παρακαλούμε λοιπόν τη γαλλική καμπίνα να μιλάει λίγο πιο δυνατά. Ωστόσο, πολύ σπάνια οι Γάλλοι είναι χαμηλόφωνοι. Συγχωρήστε με, λέει ο πρόεδρο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, συμφωνείτε. Πρώτα έχουμε το Μνημόνιο Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα τη πολιτική αεροπορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Έτσι μπορούμε να ελέγξουμε και το σύστημα. Αρχή της ψηφοφορίας. Ωραία. 46 ε, υπέρ, ε, κανένας κατά, καμία αποχή, ε, μία αποχή. Ε, ωραία και χαίρεται ο εισηγητής. Περνάμε στο σημείο 12, το οποίο είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Έχουμε εδώ την έκθεση της κυρίας ε, Ματίας ε, με πολλές ε, τροπολογίες. Ξεκινώ με τον συμβιβασμό υπαριθμών 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές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 κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 154 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.96 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Η κυρία Ματία θέλει το λόγο. Όχι. 296 ε. με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ. «306 έχουμε προφορική τροπολογία». Δεν την έχω όμως. Έχετε την προφορική τροπολογία το 306. Κύριε Ματίας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όντως υπάρχει μια προφορική τροπολογία που θα ήθελα να τη διαβάσω στα αγγλικά. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε ε, το συνολικό κόστος ε, του ορίζοντα 2020 θα αναθεωρηθεί. Ζητάει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει το ποσοστό που ε, αφορά το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και ζητά την διατήρηση του ποσοστού στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Θέλει κανείς το λόγο για αυτή την τροπολογία? Όχι. Τότε μπορούμε να ψηφίσουμε 306 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 το συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 324 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ, κατά, Να, να το ξαναδώ παρακαλώ αυτό. 326 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. 341, ε, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 347 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 349 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 360 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 366 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 367 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 378 υπέρ. Κατά. Να το, δω, να το ξαναδώ αυτό παρακαλώ. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, φτάνουμε στην 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή ΦΕΜ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 14 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 18 χωριστή ψηφορία το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θες 14 το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 4 το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτά. Ε, τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. And the vote. One. One EPP too many. One EPP too much. Hello, help me. Έχουμε μία ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚ. And now, and the vote is closed. Καλύτερα τώρα, ωραία, λήξη της ψηφοφορίας. με σαφή ε, πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Ματίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και όσους συνεργάστηκαν, ε, τους κοιόδης εισηγητές ε, και άλλους. με τους συμβιβασμούς είναι κάπως πιο εύκολη η ζωή μας κατά τη ψηφοφορία. Κυρία Ματίας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα τα έκανα υπό κανονικέ συνθήκε, αλλά κατ' εξαίρεση θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους διέκοψαν τις θερινές τους διακοπές για να συνεργαστούν μαζί μου και να συνεχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σουζάννα και τον Αλβέη Άραν για την προσήλωση, την αφοσίωση, τον ε,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 αποχές εγκρίνεται. 9 ε, σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 11. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, Παρακαλώ να το ξαναδώ αυτό. Το δεύτερο μέρος της 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε καλύτερα. ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. 11. Το δεύτερο μέρος. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε.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 Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κάτι ξέχασα. Ε, την 21 πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα την 23 όμως, ε. Και την 22 πρέπει να ψηφίσουμε. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 32 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές εγκρίνεται 34 και 35 είναι όμοιες ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Καταπίπτουν εφόσον εγκριθεί η 34-35. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά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 Αρχή της ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έχει και πάλι μια ψήφο παραπάνω. Μα τι γίνεται. Κάτι έγινε μετά τις διακοπές. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Τζαβέλα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέρφους. Σας ευχαριστούμε για τις εργασίες σας στο θέμα αυτό. Περνάμε στην έκθεση Beauty Coffer. Ο συνάδελφος Τούρμες θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπιτικόφερ δεν μπορεί να είναι παρόν. Ε, ε, ε μου ζήτησε στη θέση του να ευχαριστήσω τους κύριους συζητές για την ε, πολύ καλή συνεργασία. Αν ψηφίσουμε, επειδή θα ψηφίσουμε και για τον ε, αντιδραστήρα ΙΤΕΡ, ως ε, πράσινη ε, είμαστε κατά, του, ε, κατά της πυρηνικής ενέργειας. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν θα πρέπει να δώσουμε τόσα χρήματα για το θέμα αυτό. Πάντως ο εισηγητής με, με τον σκιώδη εισηγητή γενικά ήταν ικανοποιημένος με τα υπόλοιπα μέρη. τα σημειώνουμε αυτό στα πρακτικά και προχωράμε στην ψηφοφορία. Είναι πλοκή τώρα η ψηφοφορία. Τα νούμερα λέω. υπέρ. Κατά. 6088 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Να ελέγξουμε. 60-88 την ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για την 60 Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δίκιο είχα. Τα δύο τελευταία νούμερα θα λέω, συμφωνείτε. 25. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Λοιπόν, υπέρ κατα Αποχέ Αποχές εγκρίνεται. 0-0. Όχι, δεν την ψηφίζουμε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 01, υπέρ, 61, 01. μηδέν ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 15 είναι όμοια 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 02 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 03 υπέρ κατά αποχές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 Να την ελέγξουμε. Εντάξει. Ελέγχουμε την 21. Υπέρ. Ε, αρχή της ψηφοφορίας, συγγνώμη. Ε, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 ε, υπέρ. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα σε χωριστή ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο και τρίτο μέρος. Δεύτερο μέρος της 24, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά. Παρακαλώ το ξαναδώ αυτό, 90 υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε, την 90, αρχή της ψηφοφορίας. Closed, abgelehnt. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνάμε στην 50, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61, συγγνώμη, 51 υπέρκατα κατά ε, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Μη ζητάτε έλεγχο προτού να έχω πει το αποτέλεσμα. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 56 καταπίπτει. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά.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 Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω. 71 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε αυτό καλύτερα. Ελέγχουμε την 71. Αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 09. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στην ε, τελική ψήφο. Αρχή της ψηφοφορίας, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Μπιτικόφερ. Ο κύριος Σίλερ, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή σας. Δεν θέλω να αφήσω ασχολία στο αυτό που είπε ο κύριος Τούρμες. Ε, πολύ δύσκολο θα είναι να περάσουμε τις θέσεις μας ε, στην ε, διαδικασία του προπολογισμού. Όταν έχουμε εισηγητές από πολιτικές ομάδες που καταλήγουν σε συμβιβασμό με άλλες πολιτικές ομάδες, Ε, αλλά καταψηφίζουμε τις ε, βασικές ε, τροπολογίε. Αυτό θα αποδυναμώσει πολύ τη διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής μας στις διαπραγματεύσεις αυτές. Στην διαδικασία του προϋπολογισμού τέτοια μεταχείριση ενός τόσο σημαντικού θέματος δεν θα είναι υπέρ μας. Αυτό που κάνανε σήμερα οι πράσινοι με τον εισηγητή τους ε, δεν είναι υπέρ μας. Ε, το σημειώνουμε, ο κύριος Τούρμες θα ήθελε να απαντήσει. Πολύ σύντομα. Το πρόγραμμα ITER, το να λάβει τόσα δισεκατομμύρια, τη στιγμή που εμείς ως Κοινοβούλιο Ε, δεν θέλουμε μια, πιο, μια θέση με περισσότερες ε, αποχρώσεις. Είδαμε στη Ιαπωνία πολλοί προμηθευτές ε, δεν ε, μπορούν ε, να λειτουργήσουν λόγω των καταστροφών. Με το τσέτ υπάρχουν προβλήματα και ακόμα και στην Γερμανία στους χριστιανοδημοκράτες υπάρχουν φωνές που αμφισβητούν το θέμα αυτό. Γι' αυτό είπαμε αυτά που είπαμε. Ωραία, τα σημειώνουμε αυτό. Σας παρακαλώ μόνο μια γενική παρατήρηση. Ο καθένας ε, και η κάθε πολιτική ομάδα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση ε, να ψηφίσει σύμφωνα με τις πεπιθήσεις του. Ε, δεύτερον, υπάρχουν φυσικά θέματα για τα οποία θα ακουστεί η φωνή μας μόνο εάν Ε, μιλάμε ενωμένοι. Αυτό είναι σωστό και σημαντικό. Θα το λάβουμε όλοι αυτό υπόψη μας, ε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, πολιτικές διαφορές, ε, δεν μπορούμε να τις ε, παραπλέψουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 15 της ημερησίας διάταξης προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη. Αν συμφωνείτε θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πατριτσέλο, διότι είναι εισηγητής. Κυρίες και κύριοι, λίγη ησυχία παρακαλώ. Κύριε Πατριτσέλο, περιμένετε σας παρακαλώ λίγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσετε το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσει να μας παρουσιάσει συνθετικά και μετά να ακολουθήσουμε εμείς σύμφωνα με τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι, προβλεπόταν να πάρει η Κομισιόν πρώτο λόγο, αλλά ήθελα για να είμαι δίκαιο να σα δώσω πρώτο λόγο. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν. Δίνω λοιπόν πρώτα το λόγο στην Κομισιόν. Ε, ποιον εκπρόσωπο έχουμε εδώ. Ο κύριο Αγκούστο Γκοντζάλε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ανακοίνωση. Καταρχήν, ο τίτλος της είναι «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη». Είναι σαφής ο τίτλος και το μήνυμα που μεταδίδει. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική θα πρέπει να είναι ένα μέσο για προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών που θα ευνοεί τους πολίτες παρά αυτό που πιστεύουν πολλοί, το διάστημα είναι κοντά στις ε, χερσαίες μας δραστηριότητες ε, και οι διαστημικές ε, στρατηγικές συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, στις μεταφορές, στην ανθρωπιστική βοήθεια και η διαστημική στρατηγική συμβάλλει στους στόχους του 2020 γιατί δημιουργεί γνώση, καινοτομία, διευρύνει την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει την ευρωπαϊκή θέση στην παγκόσμια σκηνή. Με αυτό το υπόβαθρο λοιπόν στην ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε σαφεί προτεραιότητες για την ανάμειξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα. Καταρχήν η ευόδοση του προγράμματο Γαλλέο και σε αυτά τα προγράμματα θα συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών αυξάνοντα την ασφάλεια των μεταφορών, ενισχύοντα τι υπηρεσίε προ του ε, ηλικιωμένου και του. Ε, αναπήρουσα και θα έχει ωφέλειε στις μεταφορές, την ενέργεια, την ασφάλεια, το περιβάλλον, σε πολλού τομεί τη οικονομίας δηλαδή. Δεύτερον, η παγκόσμια παρακολούθηση για το πρόγραμμα του περιβάλλοντος, GNES, που θα έχει ρόλο κλειδί για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την, των κλιματικών αλλαγών. Θα συμβάλλει στη διαχείριση των κρίσεων και υποτροπή του, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην προστασία των πολιτών, όλα αυτά τα θέματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και θα δημιουργήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες ε, με τη χρήση καλύτερης της πληροφορίας. Επίσης, ε, σε ό,τι φορά την ε, ασφάλεια στο διάστημα, τρεις είναι οι άξονες αυτής της προτεραιότητας. Καταρχήν το GNES συμβάλλει στην διαχείριση των συνόρων, υποστήριξη της εξωτερικής δράσης και παρακολούθηση των θαλασσών. Επίσης συντονίζει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση υπάρχουσας διαστημικής υποδομής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών για τη διαχείριση των κρίσεων και για την βελτίωση της ασφάλειας γενικώ. Τρίτον και πολύ σημαντικό θέμα, η προστασία της ε, διαστημικής υποδομής κατά της ηλιακής ε, ακτινοβολίας ή της σύγκρουσης. Η διαστημική υποδομή έχει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία και την ευημερία της κοινωνίας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ό,τι αφορά ε, τους διαστημικούς μας στόχους. Από οικονομική άποψη και δημοσιονομική δράση αυτές θα πρέπει να ε, διεξαχθούν στα πλαίσια των ορίων του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων τη Διαστημική Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων τη. Ο διαστημικό κλάδο, η διαστημική βιομηχανία χρήζει ιδιαίτερη προσοχή γιατί αποτελεί κλάδο κλειδί τη οικονομία μα και τη κοινωνία μα. Το 2010 ο τζίρο ήταν 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ με 35.000 ε, ιδιαίτερα εξειδικευμένε θέσει απασχόληση. Οι διορυφορικέ επικοινωνίε δημιουργούν τεράστια έσοδα και διαδραματίζουν ε, σημαντικό ρόλο και στην καθημερινότητά μας. Ε, οι δορυφόροι επικοινωνία εξασφαλίζουν πρόσβαση στο βριζονικό ίντερνετ, στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και διευκολύνουν και τι μεταφορέ. Επίσης διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας απόκριση σε περίπτωση κρίση. Οι δορυφόροι επικοινωνία ε, συμβάλλουν ε, τα μάλα και στην υλοποίηση του ψηφιακού προγράμματο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλλουν ε, στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα θα πρέπει να στηρίξει ιδιαίτερα την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών, ιδιαίτερα των τεχνολογιών που χρειάζονται για, την ανεξαρ... για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας της δαστημικής στρατηγικής και δημιουργούν πραγματικά τεχνολογικά αποτελέσματα και βρίσκονται στην αιχμή. Θέλουμε φυσικά στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για μια διαστημική βιομηχανική πολιτική. Βασική στόχη μια τέτοια πολιτική θα είναι εξορρόπηση των εξελίξεων τη βιομηχανία, συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ανάπτυξη μιας αγοράς του διαστήματος για προϊόντα και υπηρεσίες του διαστήματος. Όπως προβλέπει η ανακοίνωση, η διεθνή συνεργασία είναι ζωτική σημασία για το διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει και να ευαθύνει του ε, διαλόγου για το διάστημα με στρατηγικού εταίρου όπω είναι η ΕΠΑ, η Ρωσία και επίση ε, να, να εγκαινιάσει διαλόγου με υπάρχουσε και αναφιόμενε οικονομίε και ιδιαίτερα με την λαϊκή Κίνα θεωρούμε ότι και η Αφρική χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ώστε και η ήπειρο αυτή να επωφεληθεί από τη υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τη δορυφορική πλοήγηση και αντίστοιχε υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι και το θέμα της διαστημικής διακυβέρνησης είναι σημαντικό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία των κρατών μελών και τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε το συντονισμό και τη διαχείριση των διαστημικών προϊόντων. Ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ θερμά. Να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Πατριτσέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί παρουσίασε με συνθετικό και καθαρό τρόπο ένα θέμα αρκετά περίπλοκο, την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Νομίζω ότι η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης είναι ένα πρώτο βήμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και στον τομέα ε, της διαστημικής πολιτικής υπό το φως των στρατηγικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι φιλόδοξη γιατί οι διαστημικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας και προσθέτουν αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η σημασία λοιπόν του διαστημικού χώρου έχει υπογραμμιστεί επίσης ξεκάθαρα και από τη συνθήκη της Λισαβόνας μέσω του 189 που δίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη συντονισμού και ενίσχυσης των πολιτικών, των διαστημικών, των διαφόρων χωρών μέσω μιας κοινή στάσης που θα ευνοήσει την τεχνολογική και ανταγωνιστική πρόοδο του συγκεκριμένου τομέα. Η έκθεση της Επιτροπής μας τις επόμενες εβδομάδες θα περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προσδώσουμε αξιοπιστία στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική πρέπει να είναι αξιόπιστη και γι' αυτό πρέπει να έχει φιλόδοξους στόχους και κατάλληλη χρηματοδότηση. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ κατά πρώτον ότι είναι απαραίτητο να έχει λειτουργικά και χρηματοδοτικά μέσα επαρκή έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμόσουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις ευρωπαϊκές τύπου ΣΥΜΕΣ, γκαλιλαίο κτλ μακροπρόθεσμα και για να μπορέσουμε να υπάρξει ένα σωστός μακροπρόθεσμος προγραμματισμός είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει εγγυήσει σε επίπεδο χρηματοδότησης όχι μόνο για την αναδιάταξη των δορυφόρων που υπάρχουν αλλά για να καλυφθεί και το κόστος της τεχνολογικής τους ανάπτυξης και για να υπάρχει περιοδική αντικατάσταση αυτών που φτάνουν στο τέλος του κύκλου τους. Αυτό θα δώσει συνέχεια και στήριξη λοιπόν στα συστήματα αυτά. Είναι σαφές ότι τα διαστημικά συστήματα χάνουν τις επιδόσεις τους και ε, τον, την ανταγωνιστικότητά τους με το χρόνο απέναντι και στους ανταγωνιστές. Γι' αυτό λοιπόν και για το Γαλιλαίο το σύστημα είναι απαραίτητο για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ε, ε, διαστημικής πολιτικής να εντάσσεται στον προϋπολογισμό ε, και όχι να βρίσκεται εκτός του προϋπολογισμού γιατί κάτι τέτοιο θα υπονομεύσει την ε, επιβίωσή του. Είναι κάτι που το καταδικάζει στο μέλλον και αυτό είναι και κάτι το απαραίτητο για τον Ευρωπαίο πολίτη. Πρέπει να υπάρχει χρηματοδοτική διαθεσιμότητα λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής επιτρέποντας να υπάρξει συνέχεια στη στήριξη φιλόδοξων, φιλόδοξων συστημάτων GMS. Νομίζω ότι πέραν των χρηματοδοτικών προβλημάτων θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες εθνικές υπηρεσίες ή ευρωπαϊκές υπηρεσίες για τη διαχείριση των κοινών προγραμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε ποια είναι οι βασικές αρχές για την προστασία των διαστημικών εξοπλισμών που θα πρέπει να ενταχθούν και στα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να αποφύγουμε επιφυλάξεις, ε, επικαλύψεις συγγνώμη, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο τις υπάρχουσες υποδομές για τις οποίες τα κράτη-μέλη έχουν ε, κάνει σημαντικές επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν και η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι σημαντική για την πολιτική τη διαστημική και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το 189 να είναι σε θέση να δώσει εγγυήσει για την επιστημονική επιβίωση ενός χώρου όπως το διάστημα στον οποίο η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι προϋπόθεση. θα δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Κλάντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, ξεκαθάρισε τι ωφέλη θα έχουμε από την ε, διαστημική πολιτική. Αυτό φαίνεται και στο έγγραφο. Δεν θα πρέπει όμως να προδικάσουμε τα πράγματα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ευρεία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ε, τρία πράγματα θα ήθελα να ε, αναφέρω, τα οποία ε, νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε Ε, πώς θα τα ρυθμίσουμε στο μέλλον. Τα δύο από αυτά τα ε, ανέφερε η ίδια ο προλαλή και εγώ πιστεύω ότι τα κονδύλια για τον ε, τομέα αυτό θα πρέπει να αντιστοιχούν στους στόχους. Βλέπουμε συνέχεια ότι διάφορα συμβούλια, επιτροπές κτλ. θέτουν πάντα ευγενείς στόχους, δεν βλέπουμε όμως πάντα αποτελέσματα. Το δεύτερο που επίσης αναφέρθηκε όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση ε, και το GMS, ε, τον Γεωστατικό Μετρολογικό Δορυφόρο, αυτά με βρίσκουν αντίθετο. Το δεύτερο θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε στα προγράμματα αυτά να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα εκτελέσει. Όσον αφορά το σύστημα GMS Galileo, είδαμε ότι είναι καλή η συνεργασία με την ΕΣΑ, με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Υπάρχουν όμως ε, πάντα προβλήματα. Ε, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των 27 κρατών μελών μια χούφτα επιχειρήσεις ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ε, θα πρέπει όμως να πετύχουμε θέμενη αξία μέσω της διαστημικής πολιτικής. Και ένα τρίτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάποιοι συνάδελφοι τον Ιούλιο στη Ρώμη ε, είδαμε από κοντά ε, τις εγκαταστάσεις του Γαλιλαίου. Ήταν ε, πολύ ωραία εμπειρία να τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Ε, είδαμε και την ε, και τις καιροτόμες λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά κτλ. Υπάρχουν εδώ πολλά επιμέρους προϊόντα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης υπάρχει το θέμα της ε, διτής χρήσης, ε, της στρατιωτικής χρήσης δηλαδή των ε, δεδομένων από τέτοιους δορυφόρους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα οι ευρωπαϊκέ οι ευρωπαϊκές ειρηνευτικές ή άλλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν πρόβλημα με αυτό όμως. ε, πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της στρατιωτικής χρήσης και να καταστήσουμε σαφές απέναντι στους πολίτες ότι αν ε, στέλνουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε διάφορα μέρη του κόσμου ε, θα πρέπει να τους δώσουμε και τα απαραίτητα μέσα για να εκτελέσουν τις ε, αποστολές τους. Αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι θα δούμε μια πολύ καλή έκθεση στο τέλος. Ευχαριστώ, συνάδελφος Ρεμέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για πολύ καιρό αισθανόμαστε την έλλειψη μιας τέτοιας ανακοίνωσης. Δεν θέλω να επαναλάβω τα σχόλια των προλαλισσάντων. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην Ευρώπη έχουμε μια, ένα σημαντικό κληροδότημα και πλούσια τεχνογνωσία για τα θέματα αυτά. Θυμάμαι ότι υπήρχε σφοδρός ανταγωνισμός ό,τι αφορά την ε, εξερεύνηση του διαστήματος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Εγώ ζούσα και εργαζόμουν στην ανατολική πτέρυγα αυτής της αντιπαλότητας ε, και παρά αυτό το σφοδρό ανταγωνισμό, το 1995 είχαμε ένα κοινό σχέδιο για το δορυφόρο Απόλλωνα με πολλά θετικά αποτελέσματα και πλεονεκτήματα που προηγουμένως θα φαίνονταν αδιανόητα και ασύλληπτα. Και έτσι καταλήξαμε σε, στην ε, κατάρτιση ενός ε, κοινού αγγλορωσικού ε, λεξικού του διαστήματος, πολύ χρήσιμο για την διεθνή συνεργασία σε θέματα διαστήματος. Τότε η Ευρώπη ήταν σχετικά πουσα, αλλά παρόλο που δαπανούσε λιγότερα κονδύλια, δεν ε, βρέθηκε πολύ πίσω από τις ε, δύο υπερδυνάμεις και αυτό δεν εκτιμήθηκε αρκετά. Η Ευρώπη έχει αλλάξει και ο κόσμος ολόκληρος έχει αλλάξει και χαίρομαι για την στρατηγική που αναπτύσσουμε τώρα. Επίσης, ε, επικροτώ το ότι μιλούμε εδώ για το Γαλιλαίο, το Άγνος, το GMS και συμφωνώ και με τον κύριο Γκλάντε ότι η διαστημική πολιτική έχει και ένα σκέλος σημαντικό που αφορά την ασφάλεια. Και ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι ότι πολύ σωστά το έγγραφο υπογραμμίζει την ανάγκη ανεξάρτητης προσέγγισης της στρατηγικής του διαστήματος. Το θέμα του κούρου είναι πολύ σημαντικό. Γενικώ πάντως πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο διορατικό έγγραφο που θα είναι και αρκετά ελαστικό για να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και να τροποποιείται εύκολα ανάλογα με τις προκλήσεις και τις ανακαλύψεις που αναπόφευκτα θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Κοινός μας στόχος είναι μία προσγειωμένη εντό εισαγωγικών διαστημική στρατηγική που θα είναι κοντά στον πολίτη και προσιτή και οικία, ώστε να καταλάβει ο απλός πολίτης για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια διαστημική πολιτική. Για τα κονδύλια θα μιλήσω καν, είναι όντως μείζον αυτό το ζήτημα, το οικονομικό, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να διαβιβάσουμε το μήνυμα ότι αν ε, θέλουμε σήμερα να εξοικονομήσουμε κάποια εκατομμύρια, στο μέλλον θα μας λείψουν δισεκατομμύρια εξαιτία της υστέρησης που θα σημειώσουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ξεχωριστή χρηματοδότηση των σχεδίων αυτών και όχι εξάρτησή τους από άλλα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Στοσνόφσκι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα όσα ήδη υπόθηκαν. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το, το έγγραφο. Εν μέρη, επειδή περιγράφει την διαστημική υποδομή που χρειάζεται η Ευρώπη, πρόκειται για έναν τομέα όπου τα μεμόνα κράτη-μέλη θα έπρεπε να αγωνιστούν σημαντικά για να πετύχουν τη δημιουργία διαστημικής υποδομής από μόνα τους. Πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα της ε, αποτελεσματικότητα ε, του συνδυασμού ε, των προσπαθειών και της χρηματοδότησης για να μπορούμε να μοιραστούμε κατόπιν και τα ωφέλη. Σαφώς η διαστημική υποδομή Η διαστημική τεχνολογία θα μας βοηθήσει στη διαχείριση ε, άλλων τεχνολογιών ε, και συμφωνώ με τον κύριο Γκλάντε ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα με σαφείς κανόνες χρηματοδότησης, διότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί με τέτοιου είδους έργα είναι να πραγματοποιηθούν με τρόπο κατακαιρματισμένο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Και από την εμπειρία μας στο παρελθόν θα πρέπει τουλάχιστον ε, να εξάγουμε την ε, προειδοποίηση ότι θα πρέπει να φροντίσουμε το Galileo και το GMS να έχουν σωστή διαχείριση. πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ε, χρηματοδοτικής ροής. Διότι σίγουρα δεν χρειάζεται να δούμε συνέχεια της κατάστασης ε, που είδαμε μέχρι τώρα με τον Καλλιλέο. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε μια προσέγγιση πιο ισχυρή. Είναι ένα έργο το οποίο θα μας δώσει νέες τεχνολογίες για το μέλλον ε, στους τομείς της ασφαλείας ε, των μεταφορών και άλλων. Θα είναι κρίμα ε, εάν δεν δούμε ωφέλη από τα χρήματα που ήδη έχουμε δαπανίσει για τα έργα αυτά. Γι' αυτό επικροτώ την έκθεση αυτή η οποία περιγράφει την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε διότι πρέπει να αποφύγουμε κάθε είδους ε, παρανοήσεις που να αφορούν ε, είτε τη χρηματοδότηση είτε τον στόχο ε, της δημιουργίας ε, διαστημικής υποδομής. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο συνάδελφος Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνει η έκθεση του συναδέλφου Πατριτσέλο. Ε, για μια ακόμη φορά θα πρέπει να σημάνω τον κόδωμα του κινδύνου για το πρόγραμμα GMS. Ο καθένας από τους συναδέλφους υπογράφησε τη μεγάλη σημασία που έχει το GMS για όλους μας. Το βασικό πρόβλημα είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Μέχρι τώρα πάνω από 3 δις ευρώ έχουν επενδυθεί στο GMS μέσω της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θεωρούν ότι τα χρήματα αυτά δαπανήθησαν σωστά. Παρόλα αυτά και εξεπλάγημεν γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 29 Ιουνίου να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα GMS εκτός του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και να αφήσει στα κράτη-μέλη την επιλογή του ύψους της συμμετοχής τους. Η πρόταση αυτή είναι μία μείζων απειλή για τη διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θέτει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό στον κόσμο πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγέτιδα στον κόσμο στον τομέα της γεωδεσικής παρατήρησης και της ε, προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρωπιστικής προστασίας. Αντίθετα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα GMS, σαν δεύτερο πρόγραμμα φάρος της Ένωσης για το διάστημα, θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται αντικείμενο χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό γιατί αλλιώς κινδυνεύει να διαλυθεί σταδιακά. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα. Στα πλαίσια αυτού του πλαισίου κρίσης, τα κράτη-μέλη έχουν ενταχθεί σε ένα αγώνα προς τη λιτότητα και την δημοσιονομική αυστηρότητα και αναπόφευκτα θα υπάρξει μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πλέον αλλά κάρτα. Μια ξεκάθαρη ανάληψη υποχρέωσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη. Η επανένταξη λοιπόν του GMS στο μελλοντικό δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο επί τη βάση των ποσών που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 834 εκατομμύρια κατέτος δηλαδή, είναι κάτι το απαραίτητο. Και ζητώ από τον ε, εισηγητή μας που είναι και η θέση του να καταστήσει το σημείο αυτό βασικό στο έγγραφό του και όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε το GMS να διατηρηθεί στα πλαίσια τα δημοσιονομικά. Νιμπλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά και πολλούς ε, συναδέρφους ε, που ήδη αναφέρθηκαν στο θέμα της χρηματοδότησης ε, του GMS. Θα ήθελα να επικεντρώσω την παρέμβασή μου στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την Κομισιόν. Στην ανακοίνωση, όπως είπαν οι συνάδελφοι, αναφέρεται ότι προβλέπεται η χρηματοδότηση του GMS από το 2014 μέχρι το 2020. Ωστόσο γράφει ότι ε, το GMS θα πρέπει να είναι ένα μέτρο που θα έχει προτεραιότητα. Εφόσον η Κομισιόν θέλει να έχει μια συνεπή πολιτική, πώς ε, μπορεί Πώ μπορεί η Κομισιόν να λέει ότι έχει προτεραιότητα αυτό χωρί να έχει διασφαλιστεί απόλυτα η ε, χρηματοδότηση. Οι συνάδελφοι ανέφεραν ότι εδώ δεν αγωνιζόμαστε κατά της Κομισιόν. Ε, κανονικά θα πρέπει να επιδιώκει τους ίδιους στόχους με ε, το Κοινοβούλιο. Ε, γρήγορη εκτέλεση, δηλαδή γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος ε, Galileo GMS ε, και γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς μπορεί να υπάρχει τέτοια συνέπεια στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Θα ήμουν ευγνώμων εάν ο πρόσωπος της Κομισιόν θα μπορούσε να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό ε, να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στην Κομισιόν για να απαντήσει. Παρακαλώ κύριε Κοντζάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρίσκει να υπάρχει κάποια αντίφαση ανάμεσα στον τρόπο που η ίδια παρουσίασε τη χρηματοδότηση του GMS στην ανακοίνωσή της και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο υποχρέωσή μας είναι να χρηματοδοτήσουμε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναγνωρίζει την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στον Καλλιλέο και το GMS, αλλά κάνει μια διάκριση ανάμεσα στα δύο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του Καλλιλέου. Προσπαθεί να συνδυάσει λοιπόν την ανάγκη χρηματοδότησης που υπάρχει στο εσωτερικό των περιορισμών που ισχύουν για όλες τις κοινοτικές πολιτικές και ταυτόχρονα να υπάρξει και η προτεραιότητα για το GMS και γι' αυτό ακριβώς ε, βλέπετε το τι λέμε για το GMS και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς αναζητήσαμε ένα αλλακτικό τρόπο για τη μελλοντική χρηματοδότηση του GMS εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού. Είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για τη μελλοντική χρηματοδότηση του GMS. Ε, τα πρακτικά θέματα θα ρυθμιστούν εν την Ωραία, σημειώνουμε αυτά που μας είπατε. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση. Ε, Απευθύνομαι και προς την Κομισιόν φυσικά. Νομίζω ότι ο κύριος Γκλάντε είπε ότι ε, η διαστημική πολιτική σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας είναι ένα από τα σημαντικά έργα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να ε, διατεθούν και τα απαραίτητα κονδύλια και για τα προγράμματα που ήδη έχουν ξεκινήσει και για τα νέα που προβλέπονται. Ε, δεν ε, βοηθάει την αξιοπιστία εάν ε, προβλέπει κανείς ένα σωρό μεγάλα προγράμματα, τα οποία όμως δεν μπορεί τελικά να πραγματοποιήσει λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν με μία τέτοια διαδικασία να μην προβλέπουμε σημαντικά νέα προγράμματα χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και το είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό και όσον αφορά τις δυνατότητες ε, που θα δώσει ε, στον βιομηχανικό τομέα. Αυτή ήταν απλά μια μικρή ε, συμπληρωματική παρατήρηση. Να ξαναδώσω το λόγο στον ε, κύριο Πατριτσέλο. Παρακαλώ. Εγώ για λόγους σύνθεσης ε, κατέθεσα κάποιες, κάποια πρώτα σχόλια για το έγγραφο το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφές ότι η προτεραιότητα του GMS και η διατήρησή του στο εσωτερικό του κοινοτικού προϋπολογισμού παραμένει μια προτεραιότητα, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την πρόταση αυτή, η οποία θα γίνει αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης ε, στις επόμενες εβδομάδες. Θα το συζητήσουμε. Το θέμα θα το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταξύ μας έτσι ώστε να βρούμε μία λύση, μία λύση η οποία να είναι όσο περισσότερο αποδεκτή γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι με τους συναδέλφους θα συζητήσουμε εκ νέου το θέμα έτσι ώστε να προωθήσουμε ένα πολύ σημαντικό για την Ένωση θέμα και γενικότερα για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν το θέμα αυτό να μην είναι απλά ένα θέμα για κάποιους εμπειρογνώμονες από εμά, θα πρέπει να είναι γενικά ένα θέμα της Επιτροπής μας. Ήθελα να το πω αυτό. Δεν έχω βέβαια δικαίωμα να το πω αυτό ως πρόεδρος, αλλά... Όταν βλέπω τις ε, συζητήσεις που έχουμε εδώ στην Επιτροπή, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα θέματα αυτά. Δεν πρέπει να ε, ε, περιοριστούμε σε θέματα αλλαγής του κλίματος ε, και περιβάλλοντος. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους που το ανέφεραν αυτό σήμερα. Και περνάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, στις μεταφορές. Συνάδελφος Κάρινς έχει ασχοληθεί με το θέμα και γι' αυτό ε, δίνω το λόγο για το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσει την γνωμοδότηση προς την έκθεση Επιτροπής Μεταφορών για τη Λευκή Βήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών και ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός γιατί έχουμε κουραστεί, ήταν αρκετά παρατεταμένη συνεδρίαση. Καταρχήν, οι στόχοι της Λευκής Βίβλου μας βρίσκουν σύμφωνος. Δεύτερον, ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι φορά τις ενεργειακά αποδοτικές πολιτικές και την εξοικονόμηση ενέργειας, θα πρέπει αυτές να μην αποβαίνουν εις βάρος της κινητικότητας και επίσης θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση όλων των μέτρων ανάλογα με την ε, επίδραση που θα έχουν στην ανταγωνιστικότητα. Δεν θα πρέπει ε, λόγω της μεγαλύτερης εξοικονόμησης να χάσουμε σε ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά ε, το ρόλο του ICT, νομίζω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος των, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε ό,τι αφορά τη διατροπικότητα κάτι που ε, φτάνει με πλοίο, σε λιμάνι, μετά χρησιμοποιεί σιδηρόδρομο, οδικές μεταφορές κλπ. Η διατροπικότητα είναι σημαντική και νομίζω ότι θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα μειώσει και τις ε, απώλειες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό των ICT, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι μεγάλες οι δυνατότητές τους και μπορούν να συμβάλλουν και στη μείωση της ανάγκης ε, ορισμένων ε, ε, προβλημάτων. Επίσης θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και την αποδοτικότητα της ενέργειας. Αυτό είναι σημαντικό. Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να λάβουν σάρκα και οστά, να εφαρμοστούν στην εμπορική πραγματικότητα. Καλή η σύλληψη και ο σχεδιασμό, αλλά η εκτέλεση και εφαρμογή είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και σημείο 5, τα βιοκαύσιμα. Είναι τεράστιο το δυναμικό της αυξανόμενης χρήσης των βιοκαυσίμων που θα μειώσει την εξάρτησή μας από αλλοδαπό πετρέλαιο και παράγωγα προϊόντα του πετρελαίου. Αλλά η μεγαλύτερη ε, συμμετοχή των βιοκαυσίμων στο ενεργειακό μείγμα θα πρέπει να γίνει μετά από σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Γιατί στην πατρίδα μου, για παράδειγμα, οι συμπολίτε μου ε, έχουν μεγάλη ανησυχία σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη χρήση των βιοκαυσίμων και την επιρροή που θα έχουν στους ε, κινητήρες μια αυξανόμενη παρουσία του βιοκαυσίμου θα πρέπει να συνοδευτεί από σωστή εξήγηση και προβολή τους πολίτες ώστε όλοι να καταλάβουν την ανάγκη χρήση τους. Αυτά είναι τα πέντε σύντομα σημεία της γνωμοδοτησής μου και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κάρινς γιατί ήταν πολύ μεστή η γνωμοδότησή του. Εγώ θα ήθελα να μείνω στα σημεία 2 και 5 των προτάσεών του. Συμφωνώ και χαίρομαι που ανέφερα ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης της ενέργειας δεν θα πρέπει να είναι αντιφατικές με το στόχο της ανταγωνιστικότητας, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούν η μία πολιτική την άλλη. Υπάρχουν πολλέ αποδείξει άλλωστε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει στην αύξηση του ανταγωνιστικότητα και όχι το αντίθετο και μάλιστα το επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που για την ε, διάρκεια ζωή ενό ε, φορτηγού ε, δείχνει πόσο η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να ε, παρατείνει το, το χρόνο χρήσης του φορτηγού και χρειάζονται περίπου 4 χρόνια για την απόσβεση του αρχικού κόστους ε, επένδυσης εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η απόσβεση αυτή γίνεται και η ανταγωνιστικότητα αυξάνεται. Άλλωστε, όλα, όλες αυτές οι τεχνολογίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα των μεταφορών ήδη ε, υπάρχουν στην αγορά, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τίποτα καινούριο, ήδη υπάρχουν και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Άλλωστε, ε, ήδη είχε αλλάξει και η συμπεριφορά των καταναλωτών. Στην πατρίδα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ο αριθμό των ε, οχημάτων ε, που παράγουν λιγότερο από 100 γραμμάρια διοξιδίου του άθρακα ένα χιλιόμετρο, και αγορά τέτοιων αυτοκινήτων έχει διπλασιαστεί. Το 2010 είχαμε 50.000 τέτοια αυτοκίνητα. Οι ίδιοι καταναλωτές δηλαδή καταλαβαίνουν ότι με την εξοικονόμηση ενέργεια εξοικονομούν και χρήματα. Σε ό,τι αφορά το σημείο 5, Χαίρομαι που αναφέρατε την αυξημένη αναλογία των βιώσιμων βιοκαυσίμων. Είναι πολύ σημαντικό τα βιοκαύσιμα να είναι βιώσιμα και να δούμε τι συνιστά βιώσιμο βιοκαύσιμο και τι όχι. Και αυτό το σημείο είναι σημαντικό για φορά, σε ό,τι αφορά την ε, ε, χρήση γης για την ε, καλλιέργεια δημητριακών που θα δώσουν βιοκαύσιμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα μη βιώσιμα βιοκαύσιμα. Αλλιώς δεν έχει νόημα η συμπερίληψή τους στο μείγμα, η αύξησή τους. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές βιοεθανόλης από τη Βραζιλία, έχουμε ένα φάσμα βιοκαυσίμων που έχουν αποδείξει τη βιωσιμότητά τους και δικαιολογούν την αλλαγή της χρήσης γης, αλλά δεν ισχύει για όλα. Επίσης, έχουμε μεγάλο δυναμικό στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έχουμε ε, βάσιμα επιχειρήματα ότι μπορούμε να παράγουμε βιώσιμα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Και υπάρχει διαδικασία διαπαιδαγώγησης, εξήγησης, ώστε να αισθάνονται και οι καταναλωτές άνετα με τη χρήση τέτοιων καυσίμων. Ευχαριστώ κύριος Γκλάντε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, ε, ε, θα ήθελα να δώσω την εκτίμηση της σκιώσης συγγήτριας που δεν μπορεί να είναι παρούσα η κυρία Τόμσεν. Πιστεύει ότι εδώ αναφέρονται πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ωστόσο λείπει κάτι πολύ σημαντικό, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός ε, μέλλοντος απειλαγμένου από ε, διοξίδιο του άνθρακα είναι, διοξίδιο του άνθρακα είναι ακριβώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, από πού θα βρούμε την ενέργεια για να φορτίσουμε τα αυτοκίνητα αυτά, τι γίνεται με το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, της δέσμευσης ενέργειας και θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στα θέματα αυτά. Η κυρία Τόμσεν θα υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Αυτά από την κυρία Τόμσεν ε, και μια προσωπική δική μου παρατήρηση. Ε, ο εισηγητής αναφέρθηκε στα εναλλακτικά καύσιμα και την αποδοχή τους από τους πολίτες. Προέρχομαι από μεγάλο κράτος μέλος όπου υπάρχει και εδώ πρόβλημα με την μίξη με αλκοόλ. Ε, είναι πολλοί οδηγοί που φοβούνται για τα αυτοκίνητά τους ε, με την πρόσμιξη ε, αλκοόλης και έχουμε καλέσει τον σχετικό τομέα να πληροφορήσει καλύτερα το κοινό σχετικά με τα θέματα αυτά. Μάλιστα, πολύ καλά. Ο συνάδελφος Βέμπερ. Euh, Η λευκή αυτή είναι ένα πολύ φιλόδοξο έγγραφο, υπερβολικά ίσως φιλόδοξο. Να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά κείμενα κανένας από τους βασικούς στόχους της προηγούμενης έκθεσης, της ε, Λευκής Βίβλου του 2001 δηλαδή, δεν επετέφθη. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα έπρεπε κάποιοι φιλόδοξοι μακροπρόθεσμα στόχοι να τεθούν σε μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ορίζοντα έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να δώσουν ένα πιο συγκεκριμένο προσανατολισμό στις δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν. Οι μεταφορές του αύριο θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες για κινητικότητα των πολιτών και στην σωστή, θα έλεγα, περαίωση των οικονομικών συναλλαγών. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να, ε, για με περισσότερο ομαδικές μεταφορές και ε, προσφυγής επίσης τεχνολογιών οι οποίες βοηθούν την κίνηση των αυτοκινήτων μειώνοντάς την αν αυτό είναι δυνατόν ιδιαίτερα για το χώρο της εργασίας. Λυπάμαι λοιπόν που στο κείμενο αυτό η κινητικότητα και η προσβασιμότητα όπως και η θεμελιώδης έννοια της εδαφικής συνοχής των τομέα των μεταφορών είναι ανεπαρκώς ε, αντιμετωπίσιμη ένα ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών δεν θα μπορέσει να υπάρξει χωρίς σαφέστατη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στο έδαφος. Να υπογραμμίσω επίσης ότι αυτή η λευκή βίβλος περιλαμβάνει σε ένα της τμήμα ε, μια έκκληση, ένα προσπάθεια καθορίζοντας δέκα συγκεκριμένους και αριθμητικά προσδιορίσιμους στόχους Νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια αυτή. Η ένατη, ο ένατος αυτός στόχος έχει σημασία, αλλά σε αυτόν δεν υπάρχει αριθμητικός ή ποσοτικός προλογισμός. Λέγεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί περισσότερο το σύστημα χρήστης ε, αυτός που πληρώνει και ε, ε, αυτός που μολύνει επίσης πληρώνει. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει πιο συγκεκριμένη ε, παρουσίαση της βασικής αρχής του όποιος μολύνει πληρώνει και να δούμε αν θα πρέπει να υπάρξει επιβολή φόρων στις οδικές μεταφορές, στις αερομεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές, κάτι το οποίο ίσως να μείωνε και τον ελκυστικό τους χαρακτήρα. Να ρωτήσω αν ε, υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν που θέλει να πάρει το λόγο. Ωραία, ο κύριος Κάριν τότε και πάλι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Τότε μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και να σας πω ότι ε, προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι ε, η 7η Σεπτεμβρίου. Ναι. Εάν θέλει κανείς να υποβάλει τροπολογίες θα πρέπει να έχει γίνει αυτό μέχρι τότε και ο κύριος Κάρινς ε, θα εργαστεί για να βρει ε, κάποια λύση. Ωραία, κλείνουμε το θέμα αυτό στο σημείο 17 δεν έχω να πω τίποτα. Ε, ούτως ή άλλως γνωρίζετε όλοι ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 8 Σεπτεμβρίου. Ε, καλημέρα σας εύχομαι. Α, όχι, ο κύριος Οντή το λόγο, παρακαλώ. Στην αρχή της εβδομάδας ένας ευρωβουλευτής ρώτησε αν στις 8 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε. Ζητήσατε συμπληρωματικές πληροφορίες, γιατί κάποια κόμματα, κάποιες πολιτικές ομάδες, μεταξύ άλλων και δική μου, σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αποστολές. Θα γίνει ψηφοφορία στις 8 Σεπτεμβρίου ή όχι. Κοιτώ τη γραμματεία μου λέει ναι. Εντάξει. Θα πρέπει να γίνει σχετική συνεννόηση. Δεν είναι πολύ καλή η λύση αυτή, απαραίτητη όμως. Αν μπορούμε να το αποφύγουμε, θα το αποφύγουμε, θα το εξετάσουμε. Ε, υπάρχουν όμως πράγματα για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις εντός κάποιων προθεσμιών. Θα ήθελα να ενημερωθούμε το συντομότερο δυνατόν, παρακαλώ. Auf Wiedersehen, das war's für heute. Σας χαιρετώ, τελειώσαμε για σήμερα.